Κέιρα Λέιλα Εταέμπ που έχουν λάβει θέση στα επίσημα θεωρία. Η εν λόγω αντιπροσωπεία πραγματοποιεί τις ημέρες αυτές επίσκεψη εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την 10η Διακοινοβουλευτική Συνάντηση Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο-Κοινοβούλιο Αλγερίας η κυρία Εταέμπ, η οποία είναι πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Κατάρτισης, Ανώτατης Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και Θρησκευτικών Υποθέσεων του Συμβουλίου του Έθνους της Αλγερίας και ο κύριος Πιέρ Αντώνιο Παντσέρη, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ, προείδρευσαν από κοινού στην ελόγω συνεδρίαση. Ελπίζω ότι οι συναντήσεις που είχατε στο Ευρωκοινοβούλιο, αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν αποδοτικέ και ότι θα συμβάλλουν ενεργά στην προσέγγιση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία τη της τη κυρία κυρίας Μάθιου σχετικά με την απαλλαγή οικονομικό έτους 2008 το European Police Academy. Τον λόγο έχει η συγγήτρια η κυρία Μάθιου. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι,